El señor presidente. Señorías, se abre la sesión. Ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Παρακαλώ πολύ καθίστε. El acta τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης σας διανεμήθηκαν. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, ε, τα θεω, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Sí, señora Harms. Κυρία Χάρμς. ¿Ha τη usted la Χάρμς. Έχετε ζητήσει το λόγο, κύριε Χάρμς. Όχι για τα χτεσινά πρακτικά, Πρόεδρε. Eh, Από την ε, ομάδα του Λαϊκού Κόμματος έχουμε πάρει τις εξής τροποποιήσεις στους ε, διορισμούς ε, μελών σε επιτροπές. Επιτροπή Αναφορών. Η κυρία Ματσόνη αντικαθιστά την κυρία Γκαρντίνη στην Επιτροπή Οικονομικών ε, Μεταφορών. Η κυρία Ντεβεϊράκ αντικαθιστά τον κύριο Ρικέ. Από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών έχουμε λάβει τους εξής διορισμούς για τις κοινωνικές επιτροπές. Επιτροπή Αναφορών, οι κύριοι Καμίνσκι και Κίρκχοπ. Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η κυρία Τσεσκόβα. Επιτροπή α, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο κύριος Χέλμερ. Επιτροπή Ελευθεριών, ο κύριος Μακμίλαν Σκότ. Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας, ο κύριος Κίρκχοπ. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Ντέβα και η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, ο κ. Λεγκούτκο. Περνάμε στις ε, προτάσεις ε, ορισμού μελών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Δεν έχει υποβληθεί καμία τροποποίηση, καμία αλλαγή. Συνεπώς, ε, θεωρώ εγκεκριμένες τις προτάσεις της διάσκεψης των πρόεδρων. Σενιόρα Χάρμς, κύριο usted παράβρα. Κύριε Χάρμς, έχει το λόγο. Ja, Herr Präsident. Κύριε Πρόεδρε, εχθές ε, μας ήρθε μια πολύ δυσάρεση είδηση, συγκεκριμένα από τον Κρόσνευ, από την Τσετσενία. Συγκεκριμένα, μια δημοσιογράφος ε, η Ναστάλια Ισχυμύροβα που είναι πολύ γνωστή σε εμά, δολοφονήθηκε